ε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, στην, ε, στα θεωρία των επισκεπτών. Εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια εξελίσσεται μια σιωπηρή επανάσταση πάνω στα ερήπια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Ορθώθηκε ένα μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας οικοδόμημα. Οι εχθροί έδωσαν ο ένας το χέρι στον άλλον σε ένδειξη συμφιλίωσης και οι περιοχές που είχε πλήξει ο λοιμός και η καταστροφή ενώθηκαν σε μια ιστορική αγορά, στην πρώτη ιστορική αγορά του κόσμου, απελευθερώθηκαν από δικτατορίες οι λαοί, μετετράπηκαν σε αστικές δημοκρατίες και προώθησαν ένα προοδευτικό κοινωνικό μοντέλο που όμοιο του δεν έχει στον κόσμο. Από κοινού δημιουργήσαμε ένα κοινωνικό πρότυπο, ένα κοινωνικό μοντέλο που μας επιτρέπει κάθε μέρα να ζούμε λίγο καλύτερα ένας μαζί με τον άλλον. Ένα μοντέλο της δημοκρατίας, ένα μοντέλο της ειρήνης, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης που μας συνδέει τον ένα με τον άλλον άρρηκτα και κατά τρόπο ιδιάζοντα. Πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το μοντέλο, να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αξίες γνωρίζοντας από πού ερχόμαστε και πού έχουμε φτάσει. Μέσα σε 60 χρόνια δεν ξανά έγινε πόλεμος. Άντρες, γυναίκες που είχαν ζήσει σε μία ανθρώπινη γενιά δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους που δεν είχαν μπορέσει ακόμα να ξεφύγουν από τα συντρίμια, που δεν είχαν ακόμα αρχίσει να ξαναχτίσουν τα σπίτια τους, μπόρεσαν κατά τρόπο σχεδόν σουρεαλιστικό δεδομένο των συνθηκών μέσα στις οποίες ζούσαν, να προχωρήσουν σε μία ιδέα μοναδική που θα τους επέτρεπε να αποτρέψουν τέτοιες καταστροφές στο μέλλον στην Ευρώπη. Και έτσι ξεκίνησαν μία σιωπηρή επανάσταση. Να μην ορθώνουν πια τύχη, αλλά να ανοίγουν γέφυρες συμφιλίωσης. Να μην στοχεύουν στον εχθρό, αλλά να του απλώνουν το χέρι. <coughs> να μην κατηγορούν και καταδικάζουν στον αιώνα τον άπαντα τον υπέτειο, αλλά να τον συγχωρούν. Να ανοίγουν τους φράχτες αντί να ορθώνουν τύχη. Να επιλέγουν ανοιχτή οικονομία και όχι προστατευτισμό. Ελεύθερη οικονομία και από κοινού να χαράξουν έτσι το δρόμο για την ευημερία των πάντων. Αυτό ήταν ο στόχος των ανδρών και των γυναικών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, ο Ρομπέρ Σουμάν πριν από 62 ακριβώς ημέρες, ε, χρόνια ανακήρυξε σαν σήμερα την ημέρα της αλληλεγγύης, το δρόμο για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη αυτή, η ουσιαστική αλληλεγγύη, αποτελεί και το μοναδικό δρόμο που μας υποχρεώνει να πάρουμε, εάν θέλουμε να επιβιώσουμε και εννοώ κυριολεκτικά να επιβιώσουμε και μας σε εκ τούτου να δράσουμε από κοινού, να κοιτάμε όχι μόνο τα δικά μας συμφέροντα, γιατί αυτά είναι αναπόσπαστα και ανα... Ε, άρρηκτα συνδεδεμένα με τα συμφέροντα του γείτονά μας. Να είμαστε όλοι μαζί πιο ισχυροί και όχι να προσπαθούμε ο καθένας να είναι πιο ισχυρός από μόνος του. Έτσι λοιπόν, ένα χωρίς προηγούμενο μοντέλο εδώ και έξι δεκαετίες προσφέρει στην Ευρώπη ειρήνη, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, ευημερία και αλληλεγγύη. Το πνεύμα αυτό των ιδρυτικών στελεχών, των ιδρυτών, ανδρών και γυναικών της Ευρώπης έχει μπορέσει να δώσει μέσα από τα συντρίμια απάντηση στα προβλήματα. Αυτό το θάρρος που επέδειξαν και η απάντηση που ήταν μόνο μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, μόνο μαζί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δεινά, μας αναγκάζει και σήμερα, δεδομένης και της μεγάλης οικονομικής κρίσης, της αυξανόμενης αναργίας, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, να προχωρήσουμε σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μένα αλλά που μπορούμε πολύ πιο εύκολα σε ένα μονοπάτι πολύ πιο ομαλό από αυτό που χρειάστηκε να πάρουν οι ιδρυτές πατέρες της Ευρώπης για να βρούμε κοινέ λύσεις. Κυρίες και κύριοι. Οι πρώτοι ιδρυτές της Ευρώπης ζούσαν στα ερήπια και έχτισαν την Ευρώπη. Έχτισαν μια Ευρώπη ενώ σε μεγάλο βαθμό λιμοκτονούσαν. Έχτισαν μια Ευρώπη, ενώ είχαν χάσει του, τα μέλη της οικογένειάς τους, ήταν χείρες και ορφανά, ενώ επέστρεφαν μόλις από στρατόπεδα συγκεντρώσεως όπου είχαν υποστεί βασανιστήρια και δεινά. Και όμως μπόρεσαν να δείξουν το θάρρος και να πούνε από μαζί θα τα καταφέρουμε, παρότι είχαν μια τέτοια φρικτή και αποτρόπαιη ιστορία πίσω τους αφήσει. Γιατί λοιπόν εμείς να μην μπορούμε να προχωρήσουμε πιο, με συνθήκες πολύ πιο ομαλές από ότι οι πατέρες εκείνοι που ξεκίνησαν την Ευρώπη. Γιατί αντί να ενωνόμαστε υπάρχουν τώρα κεντρομόλες δυνάμεις που, ε, που ξεχωρίζουν τον έναν από τον άλλον. Γιατί υπάρχει κίνδυνος τόσο για το ευρώ όσο και για την ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων. Τι πιο πολύτιμο έχει να μας προσφέρει η Ευρώπη από την ελεύθερη δυνατότητα να ταξιδεύουμε, να εργαζόμαστε, να εγκαθιστάμεθα σε ένα άλλο μέρος της. Η γενιά του Εράσμους που έχει ως αυτονόητο δικαίωμα να εγκατασταθεί σε ένα από το ένα μέρος στο άλλο της Ευρώπης χωρίς να χρειάζεται να περάσει τον φράχτη των συνόρων, χωρίς να χρειάζεται να δείξει διαβατήριο. Εμείς που ζούμε μέσα στο χώρο του Σέγγεν, Πώ είναι δυνατόν να ε, υποσκάπτουμε τις βασικές ιδέες τη αξία Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Κυρίες και κύριοι, δεν πρέπει να επανέλθουμε στα εθνικά σύνορα. Πρέπει από κοινού να δράσουμε για να προστατεύσουμε μαζί την, τα εξωτερικά σύνορα, την Ευρώπη, την κοινή διακυβέρνηση, το χώρο του Σέγγεν, το ευρώ. Αυτή είναι η λύση που προσφέρεται, η μόνη λύση στα προβλήματα που έχουμε. Και επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για το ευρώ. Το ευρώ είχε σαν στόχο να συνενώσει τους λαούς της Ευρώπης. Τώρα όμως έχει μετατραπεί σε σύμβολο εθνικών εγωισμών από κάθε πλευρά και κινδυνεύει να μετατραπεί σε σύμβολο του διχασμού. Μια επιστροφή όμως σε εθνικά νομίσματα θα είχε τραγικές, μοιραίες συνέπειες. Θέλουμε να αρχίσουμε να ξαναπληρώνουμε σε γερμανικά μάρκα, σε φιωρίνια, σε γαλλικά φράγκα βελγικά, φράγκα λουξεμβουριανά, φράγκα λιρέτα. δεν έχει αντιληφθεί ο κάθε ένας και η κάθε μία που βρίσκονται εδώ ότι δεν υπάρχει άλλο νόμισμα το οποίο μπορεί να επιβιώσει στον διυπηρωτικό νομισματικό ανταγωνισμό δεν θα ξεπέσουμε και πάλι εάν περάσουμε, εάν χρειαστεί να μετατρέψουμε τα αποθέματά μας τα νομισματικά, σε εθνικά νομίσματα, σε έναν διακρατικό ανταγωνισμό μικρόψυχο και καταστροφικό για όλους. Κυρίε και κύριοι, εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεκδικούμε εδώ και πολύ καιρό δημοσιονομική πειθαρχία. Αλλά το Κοινοβούλιο επίσης εδώ και πολύ καιρό διεκδικεί ένα σύμφωνο ανάπτυξης. Εάν κοιτάξουμε την κατάσταση των εθνικών οικονομιών που παρασύρονται μέσα στον κικαιώνα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης βλέπουμε ότι η οικονομική κατάρρευση της Ευρώπης και η, η αυξανόμενη ανεργία Μόνο με την ανάπτυξη μπορούν να αντιμετωπιστούν. Εδώ και πολύ καιρό ζητούμε ναι, ισοσκελισμένου προπολογισμού. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το απαιτούμε ξεκάθαρα γιατί είναι απαραίτητο. Και πρέπει να σα πω όμω, κυρίε και κύριοι, γιατί είναι βαθύτατη μου πεποίθηση ότι ισοσκελισμένο προπολογισμό είναι ταυτόχρονα και για λόγου ισότητα και δικαιοσύνη έναντι των γενεών να ε, απαραίτητος. Γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι τα δικά μου επίπεδα διαβίωσης θα ε, χρηματοδοτηθούν από τη δουλειά που θα κάνουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου μέσα σε μερικές δεκαετίες. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Και γι' αυτό χρειάζεται δημοσιονομική πειθαρχία να είναι αναμφίβολο αυτό. Ταυτόχρονα όμως λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης ότι χρειάζεται πέραν της λιτότητας να υπάρξουν πρωτοβουλίες που θα δώσουν νέα όθηση στην ανάπτυξη. Μιλούμε για ένα νέο, ίδιο πόρο, για ένα νέο πόρο ε, εσόδων των φόρων στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που έχει εγκριθεί από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου με πλειοψηφίες που δεν υπάρχουν πολύ εύκολα σε άλλα τέτοια νομοθετήματα. Έχουμε ζητήσει την πάταξη της ε, φόρου αποφυγής και φοροδιαφυγής και επιτρέψτε μου κυρίες και κύριοι να αναφερθώ πιο συγκεκριμένα ε, να αναφερθώ Στι συγκεκριμένε συνθήκε που αντιμετωπίζουμε ότι ο πραγματικό πατριώτη είναι αυτό που βοηθάει τη χώρα του να σταθεί στα πόδια τη και όχι αυτό ο οποίο κλείνεται στο καβούκι των εθνικών συνόρων, Αυτό που μιλάει για ελεγγύη. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και τη θέλουμε στα σοβαρά και η κυβέρνηση φαίνεται ότι την επιδιώκουν στα σοβαρά, δεδομένου ότι έχουν προβλέψει μια μεγάλη σύνοδο για την ανάπτυξη 23 Μαου. εάν θέλουμε να δούμε πώ θα προχωρήσουν αυτέ οι προποθέσει για την ανάπτυξη και ναι πρέπει να πούμε τι είδου μέσα και κονδύλια μας διατεθειμένα διαθέσουμε για την ανάπτυξη αυτή, τότε κυρίε και κύριοι και ως εκ τούτου κυρίες και κύριοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ημέρα που εορτάζουμε την διακήρυξη Σούμαν με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό δεν μπορεί να δέχεται προτάσεις για περικοπές του προϋπολογισμού δεν είναι καν λογικό κάτι τέτοιο. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προπολογισμό επενδύσεων. Έχει να κάνει, είναι συνδεδεμένο και με την οικονομική ανάπτυξη και με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία. Όποιο θέλει λοιπόν να φέρει την ψαλίδα των περικοπών στον ευρωπαϊκό προπολογισμό, ουσιαστικά ε, υπονομεύει το κοινό μέλλον. Σύμφωνο ανάπτυξη, κυρίε και κύριοι, μάλιστα δεν χρειάζεται κανεί περισσότερο από ότι οι νέοι στην Ευρώπη, αυτοί του οποίου απειλεί η μεγάλη οικονομική κρίση η οποία μπορεί να τους μετατρέψει σε μια χαμένη γενιά. Οι νέοι από 18 έως 30, οι νέοι της Ευρώπης, τους οποίους συνάντησα εγώ την προηγούμενη εβδομάδα στην Ισπανία. Όλοι όσοι είναι στα πανεπιστήμια, πολλές φορές έχουν και τρία πανεπιστημιακά πτυχία και είναι άνεργοι. Είναι άνεργοι χωρίς να έχουν ευθύνη για την κρίση. Πληρώνουν όμως χωρίς να έχουν ευθύνη το πολύ βαρύ αυτό τίμημα για να διασωθούν κράτη και τράπεζες. Με ρώτησε ένας νεαρός, μια νεαρή στην Μαδρίτη. Έστω να ζητήσουμε, να, να δεχθούμε 750 δισεκατομμύρια να βγουν ε, από τις τσέπες μας για να, για να σταθεροποιηθεί το σύστημα το χρηματοπιστωτικό. Αλλά εσείς ένα εκατομμύριο πότε δώσατε για εμάς τους νέους. Εμείς που θα είμαστε 20 χρόνια άνεργοι και ίσως και δεύτερη γενιά από ό,τι προβλέπεται σε ορισμένες χώρες να περάσει το φάσμα της ανεργίας. Έτσι λοιπόν χρειάζονται νέε δυνατότητε. Δυνατότητε πάνω απ' όλα για κατάρτιση και οπουδήποτε διατίθενται χρήματα για την κατάρτιση είναι χρήματα καλώ τοποθετημένα. Αυτό εννοούσε ο Γομπέρ Σουμάν με την ημέρα τη αλληλεγγύη, με την Ευρώπη και την αλληλεγγύη στην ουσία στην πράξη. Εάν καταφέρουμε να διαφυλάξουμε θέσει εργασία ή να δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασία, τότε όντω υλοποιούμε στην ουσία την ε, αλληλεγγύη. Αυτό το οποίο είναι και το πρόσωπο το πραγματικό της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε για να απαλλάξουμε ή να προφυλάξουμε καλύτερα την Ευρώπη από την ε, ε, αδιαφορία, από την απώλεια κάθε σημασίας και έννοιας. Αυτό απαιτούν οι πολίτες της Ευρώπης από μας. Πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Πρέπει να τοποθετηθούμε ρητά υπέρ της αλληλεγγύης. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τους εθνικούς ε, εγωισμούς και να αφήσουμε τις, τους διαχωρισμούς μεταξύ φτωχών και πλουσίων μεταξύ εκείνων που μπορούν και εκείνων που δεν μπορούν γιατί αυτό είναι σβάρο των πάντων και πρέπει να αναγνωρίσουμε την κοινή μας ταυτότητα. Οφείλουμε, πρέπει ως Ευρωπαίοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για ολόκληρο τον κόσμο ως Ευρώπη, ως Ευρωπαίοι. Ένα χρόνο μετά την έναρξη της Αραβικής άνοιξη, οι εταίροι μα εκεί περιμένουν από εμά να τους στηρίξουμε στη διαδικασία τη μετάλλαξη. Αυτό δεν σημαίνει περισσότερη Ευρώπη. Βλέπουμε ότι το ενδιαφέρον, οι εκλογές στη Γαλλία και την Ελλάδα, το αποτέλεσμα και το αντικείμενο των συζητήσεων των προεκλογικών δείχνει πόσο πολύ οι πολίτες συνειδητοποιούν, γνωρίζουν πόσο αλληλεξαρτώμενοι είμεθα ο ένας από τον άλλον, πόσο ζωντανή και υπαρκτή είναι η Ευρώπη στην καθημερινή του ζωή, ότι το πρόβλημα του ενός μετατρέπεται και σε πρόβλημα του άλλου. Και ξέρουμε επίσης, ξέρουν οι πολίτες, ότι οι λύσεις από κοινού μόνο μπορούν να προσφερθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη στην κατάσταση που διανύει τώρα, κυρίες και κύριοι, και παρά την κατάσταση που διανύει τώρα, αποτελεί και το μοναδικό και επιτυχές τέτοιο εγχείρημα της ιστορίας της ανθρωπότητας. Ο Σούμαν μπόρεσε με το σχέδιό του και στη συνέχεια το 58 με τις συνθήκες της Ρώμης να βάλει το πρώτο λιθαράκι με μέσα στην πορεία αυτή επίση που μας έφερε σήμερα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 μέλη και με καταπληκτικές εξελίξεις η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ελλάς απέδιωξαν τις δικτατορίες που τις τυράνευαν έχουμε ανθρώπους μεταξύ μας που είχαν ενεργά αντισταθεί στα δικτατορικά καθεστώτα. Είχαμε την πτώση του τείχους του Βερολίνου την πορεία για την απελευθέρωση των κρατών που οδήγησε στην επανένωση της Ευρώπης. Η τεχνητή διέρεση της Υπήρου μας από το σιδηρούν παραπέτασμα έληξε οριστικά. Έφερε προοπτικές ενσωμάτωσης και μεταμόρφωσης των χωρών της Κεντροανατολικής Ευρώπης και ενσωμάτωση της Ευρώπη που ενίσχυσε τη σταθερότητα της Ευρώπης. Πολλοί από τους πολίτες περιμένανε ότι η προσχώρηση των χωρών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα, άλλαζε, θα άλλαζε τα κράτη-μέλη σε εκβάθρον. Και επίσης ότι τα νέα κράτη-μέλη θα βοηθούσαν τα παλιότερα κράτη-μέλη να αλλάξουν και αυτά επί το βελτίο. Φέρανε την πολιτική τους και ιστορική τους εμπειρία οι χώρες αυτές της ε, ε, προσχώρηση του 2004 και συνέβαλαν λοιπόν <clears throat> και στην συνολική ενσωμάτωση της Ευρώπης. Το είπα αυτό και το λέω εκπεφασμένα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που έχω διαδεχτεί τον ε, κύριο Μπούζεκ, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος του Κοινοβουλίου και προερχόταν από αυτές τις χώρες. Χωρίς καμιά αμφιβολία, κύριε Μπούζεκ, είμαστε μια ενωμένη ήπειρος, μια ήπειρος κοινή αντιμετώπισης και κοινή διαβίωσης. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε τη δημοκρατία, την ελευθερία, την αλληλεγγύη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους αγώνες που έχουμε διεξαγάγει κατά της καταπίεσης, τους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Το σιδερούν παραπέτασμα, οι δικτατορίες στη Νότια Ευρώπη δεν είναι απλώς καθεστώτα τα οποία κατέρευσαν κατέρευσαν χάρη στην ειρηνική διαμαρτυρία των πολιτών εναντίον ενός συστήματος το οποίο ήταν εγκληματικό στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Οι δικτατορίες αυτές κατέρευσαν από τη δράση των ανθρώπων. Οι συνάδελφοί μας λοιπόν είναι συνάδελφοι που προήθαν από αυτές τις χώρες και σήμερα στην 9η Μαΐου θα πρέπει να θυμηθούμε όλοι την αξία της ελευθερίας και της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και ιδίως όταν έχουμε το νου μας στις χώρες του αραβικού κόσμου που και αυτοί έχουν εμπνευστεί από τις δικές μας επαναστατικές ενέργειες στην Ευρώπη που οδήγησαν στη δημοκρατία και την ελευθερία. Το παράδειγμα αυτό λοιπόν θα πρέπει να το κατανοήσουμε και εμείς πόσο σημαντικό υπήρξε και να το εκτιμήσουμε κατάλληλα. Πριν από 60 χρόνια, όπω είπα, ξεκίνησε μια σιωπηρή επανάσταση, η οποία άλλαξε για πάντα τον κόσμο μας. Η Ευρώπη έδειξε ότι είναι εφικτό να έχουμε δημοκρατία, δικαιοσύνη, ελευθερία και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών της. Η σύνδεση της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης πέρα από κάθε σύνορο μεταξύ των λαών. Αυτό είναι το μοντέλο της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Ένα μοντέλο που έχει ανεξάρτητα δικαστήρια και ελεύθερο τύπο και μέσα ενημέρωσης, το οποίο παρέχει σε όλους την υγειονομική περίθαλψη, που εξασφαλίζει ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και στα επαγγέλματα για όλους. Έχει ένα μοντέλο κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, όπου βασίζεται στη δημοκρατική και συνολική συμμετοχή. Ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την ίση εκπροσώπηση όλων των πολιτών. Ένα σύστημα το οποίο πασχίζει να φτάσει τα υψηλότερα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και έχει πράγματα υψηλότερα πρότυπα σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς αυτούς. Τονίζουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει παιδική εργασία. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες καταχρηστικές μορφές εργασίας. Έχουμε φτιάξει ένα μοντέλο στο οποίο, στο οποίο το κέντρο βρίσκεται ο άνθρωπος. Αυτή είναι η κοινωνία στην οποία εγώ θέλω να ζήσω. Και πιστεύω και εσείς το ίδιο. Ελπίζω και θέλω τα παιδιά μου, τα παιδιά σας να συνεχίσουν να ζουν σε μια τέτοια κοινωνία. Η κοινωνία αυτή όμως δεν έχει καμία εγγύηση ότι μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Είμαστε υποχρεωμένοι, χρειαζόμαστε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη και το δημοκρατικό μας υπόδειγμα θα επιβιώσει σε ένα καιρό παγκοσμιοποίηση και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το υπερασπιζόμαστε. Κάθε μέρα θα πρέπει να αγωνιστούμε και πάλι για να εξασφαλίσουμε την επιβίωση αυτού του μοντέλου. Σήμερα, την ημέρα της Ευρώπης, εμείς θα πρέπει να θυμηθούμε από πού έχουμε έρθει και πού έχουμε φτάσει. Όχι για να αυτοσυγχαιρόμεθα, αλλά για να θυμηθούμε την ιστορία μας, να διατηρήσουμε και να προασπίσουμε τα κεκτημένα μας και να τα κρατήσουμε σε μια πραγματικά ισχυρή βάση για να έχουμε δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη και σταθερότητα για το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας ευχαριστώ για την έγκριση που εκφράσατε με τα χειροκρατήματά σας. Δίνω τώρα στον Γιώσεφ Τόλ από το ΕΛΚ το λόγο. κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα γιορτάζουμε τη Μέρα της Ευρώπης. Η γιορτή αυτή της 9ης Μαΐου επέχει μια ιδιαίτερη σημασία σε μια δύσκολη και ευαίσθητη στιγμή της ευρωπαϊκής οικονόμησης και στον οικονομικό τομέα αλλά κυρίως στον πολιτικό τομέα. Πολλές φορές αναφέρουμε την πρόοδο που πετύχαν οι χώρες μας μετά από την υπογραφή της δήλωσης του Ρομπέρ Σουμάν. Και όμως <clears throat> και είναι γεγονό ότι ποτέ δεν έχουμε ζήσει ένα τόσο μακρό διάστημα ειρήνης και ευημερίας. Εμείς ως Ευρωπαίοι έχουμε πληρώσει ένα υψηλό τίμημα για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ των γειτόνων μας και ημών των ίδιων. Καταλάβαμε επιτέλου την αξία της ανεκτικότητα του διαλόγου, της αλληλεγγύη που πρέπει να ξεπερνάει του εγωισμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ανάδυση των άκρων και η άνοδο του λαϊκισμού μα εγκαλεί αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μονάχα ο οι, ακραίε παρατάξει τη δεξιά αλλά και αυτέ τη αριστερά που δεν έχουν καμία θέση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε και πολλά να χάσουμε αν αγνοήσουμε αυτή την απειλή των άκρων. Πρέπει να κατανοήσουμε του κινδύνου τη δημαγωγία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι πολίτε μα έχουν απογοητευτεί και έχουν διαψευστεί οι προσδοκίε του. Πρέπει να καλύψουμε το δημοκρατικό έλλειμμα τη Ευρώπη. Η Ευρώπη διέρχεται μια δύσκολη χρονική περίοδο. Οι αποφάσει των επόμενων μηνών θα είναι αποφασιστικέ για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα των οικονομιών μα και να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή των χωρών μα. Η κρίση του, χρέους, του χρέους, οι επιθέσεις κατά του ευρώ τον τελευταίο καιρό έχουν τουλάχιστον το θετικό στοιχείο ότι μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε το πώς έχουν, διο, ε, ολιστήσει τα δημόσια οικονομικά ορισμένων χωρών της Ευρώπης εδώ και πολύ καιρό. Με το six-pack, με το εξάπτυχο, το, τα νομοθετήματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο έχουμε δείξει ότι η Ευρώπη έχει το θάρρος να αντιμετωπίσει αυτές τις ε, καταστάσεις και να προσπαθήσει να τις ε, υπερβεί. Αλλά δεν πρέπει να μειώσουμε τις προσπάθειές μας. Μέσα σε αυτή τη ε, συζήτηση μεταξύ εξυγίανσης των εθνικών οικονομικών και της ανάπτυξης θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν μονάχα τη λιτότητα και αυτοί που θέλουν μόνο την ανάπτυξη. Είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, όπως τονίζω πάρα πολύ συχνά. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε το ένα από το άλλο. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς μείωση του χρέους και ε, όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η μείωση του χρέους, τόσο πιο ισχυρή θα είναι η ανάπτυξη. Τα μέτρα υποστήριξης της ανάπτυξης δεν μπορούν να οδηγήσουν σε πρόσθετες δαπάνες, γιατί δεν έχουμε πλέον το περιθώριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι χώρες οι οποίες ε, δαπανούν τα περισσότερα χρήματα, αν δεν κάνουν μια προσπάθεια να έχουν καλύτερη διαχείριση και μειότητα, μείωση του χρέους τους, δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Πρέπει να υπάρξει το κλίμα εμπιστοσύνη για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Και όταν μιλώ για ανάπτυξη, δεν μιλώ για μια τεχνητή ανάπτυξη, μια για μια φούσκα. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να μπορέσουμε να καταφέρουμε την ανάπτυξη. Αυτό είναι να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η Ευρώπη έχει ένα ελπιδοφόρο μέλλον υπό την προϋπόθεση ότι όλοι θα επομιστούμε τις ευθύνες μας και θα πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι απαραίτητο για κάτι τέτοιο. Πρέπει να συμπληρώσουμε την ενιαία αγορά. Πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη για να συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι, να είμαστε μεταξύ των πρωτοπόρων στι οικονομίε του 21ου αιώνα. Πρέπει να μειώσουμε το διοικητικό άχθο για να απελευθερώσουμε τι δυνατότητε των μικρομεσαίων και άλλων επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο και με την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη και θα δημιουργήσουμε τι θέσει απασχόληση του μέλλοντο. Η δήλωση του Ρομπέρτ Σουμάν άνοιξε ένα νέο δρόμο για του Ευρωπαίου σήμερα περισσότερο από ποτέ είμαστε δεμένοι ημέν με τους δε. Έχουμε δεσμούς αλληλεγγύης αλλά και δεσμούς υπευθυνότητος ημέν με τους δε. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια σύγκληση στα δημοσιονομικά αλλά και επίσης και μια σύγκληση στα κοινωνικά θέματα. Αυτή η αλληλεγγύη όμως και η σύγκληση δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα παρά μόνο με τις προσπάθειες όλων και με την εξυγίανση και την σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών. Κλείνοντας, να τονίσω και πάλι. Η δήλωση του Ρομπέρ Σουμάν μα έδωσε και ένα εγχείρημα ειρήνη το οποίο επέτυχε, ευδοκίμησε. ας το τονίσουμε και αυτό. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω η αλληλεγγύη, η ευθύνη, η πεποίθηση ο ενθουσιασμός. αυτέ θα πρέπει να είναι οι βάσει του εγχειρήματο μα στο μέλλον για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντόλ. Ο συνάδελφο κύριο Σόμποντα εκ μέρου τη ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για 6 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για τι μεγάλε προκλήσει, αλλά και για την ιστορία, αλλά και για τη συνέχεια που θα δοθεί στην Ευρώπη. Υπάρχουν όμω και απογοητεύσεις. Τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα ήταν μεγάλο, σκληρό πλήγμα απογοήτευση για μα, αλλά πάνω απ' όλα είναι απογοητευμένο ο λαό στην Ελλάδα. Είναι σε απόγνωση και αυτή η απόγνωση και η αντίσταση κατά της κοινωνικής αδικίας οδήγησε στα αποτελέσματα αυτών των εκλογών. Βλέπει ο κόσμος ότι πρέπει η Ευρώπη να δώσει ένα μήνυμα ελπίδα. Υπάρχει όμως μήνυμα ελπίδας να δώσουμε. Υπάρχουν ήδη καλά δείγματα αλλαγή και ο γαλλικός πληθυσμός, ο γαλλικός λαός επέλεξε ένα πρόεδρο ο οποίος εκπροσωπεί τις, τις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θα ήθελα να συγχαρώ στα γαλλικά τον Φρανσουά Ολαόντ για την εκλογή του και να πω ότι θα τον στηρίξουμε στο δρόμο για την αλλαγή. όπως έγραψε σήμερα ο Μάρτιν Βόλφ στους Financial Times από τους Ευρωπαίους ηγέτες μόνο ο Ολόντ έχει την ευκαιρία και την ικανότητα να βγάλει την Ευρώπη από την κρίση. Αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε. Αν μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση αυτή, μπορούμε να πιστεύουμε στην επιβίωση της Ευρώπης. Επίσης, στη Γερμανία βλέπουμε άλλες ε, εξελίξεις. Ε, δεν υπάρχει τώρα μόνο η γερμανική γλώσσα, υπάρχει και η γαλλική γλώσσα που ακούγεται ισχυρά στην Ευρώπη και ίσως αλληδημοκρατική επίσης αγαπητοί συνάδελφοι. Η μέρα της Ευρώπης σημαίνει την ανάμνηση, την ε, αναφορά στο, στην ιστορία μας, το χτίσιμο της Ευρώπης, δηλαδή πάνω στα ερήπια του Παγκοσμίου Πολέμου. Το εγχείρημα της ειρήνης. Ένα εγχείρημα ειρήνης που βρίσκεται σε κίνδυνο για άλλη μια φορά, αλλά η Ευρώπη είναι και πάνω από ένα εγχείρημα ειρήνης, είναι αυτή η οποία εξασφάλισε την κοινωνική ειρήνη στους λαούς της Ευρώπης, που στήριξε τους κοινωνικά αδύναμους και αυτή η κοινωνική ειρήνη είναι που κινδυνεύει. Γι' αυτό υπάρχουν αντιστάσεις, γι' αυτό υπάρχουν αντιδράσεις, γι' αυτό υπάρχει κοινωνική αναταραχή, γι' αυτό προτιμούν μερικές φορές οι λαοί αντιευρωπαϊκά κόμματα, κόμματα των άκρων και, και λαϊκιστικά κόμματα. Και εδώ η καταστροφή μπορεί να έχει και πολιτικό, όχι μόνο κοινωνικό χαρακτήρα. Όμως εμείς ως ελληνοδημοκράτες δεν θέλουμε πόλεμο των γενεών, δεν θέλουμε πόλεμο μεταξύ των ντόπιων και των μεταναστών. Θέλουμε μια ειρήνη, μια κοινωνική ειρήνη που θα διαφυλαχθεί και θα ανοικοδομηθεί στην Ευρώπη. Η ομάδα μου, η πολιτική, πάντοτε καθιστά σαφέ ότι ε, μέσα ότι ναι, βεβαίω ε, τα σώμεθα υπέρ μια πολιτική για την ε, δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά τα άκρα στα οποία έχει αυτή φτάσει οδηγούν σε αντίξω και μη προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Έχουμε σημαντική μείωση της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια και αντί να ασχοληθούν με την ανάπτυξη, με τι επενδύσει στην ανάπτυξη, τα κράτη, οι περιφέρειε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη ασχολούνται μόνο με περισσότερε περικοπέ στον προπολογισμό. Σα λέω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι έχει πια περάσει η κρίσιμη ώρα, έχει περάσει η δωδεκάτη ώρα. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο σε ωραία λόγια. Χρειαζόμαστε πράξεις και ουσιαστικές επενδύσεις και έναν πραγματικό νέο χρυσού κανόνα για την ανάπτυξη, για την απασχόληση μέσα από ένα δεσμευτικό βέβαια σύστημα δημοσιονομικής πειθαρχία που όμως θα προωθεί την ανάπτυξη και την απασχόληση. Δεν θέλουμε κανόνες γραμμένου σε μάρμαρο οι οποίοι έχουν αποδείξει την ιστορική τους αποτυχία. Θέλουμε ένα μοντέλο με, με ανάπτυξη και με απασχόληση. Και πάνω απ' όλα, και το αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, χρειάζονται θέσεις εργασίας για τους νέους. Πώς είναι δυνατόν να κερδίσουμε, να προξενήσουμε τον ενθουσιασμό των νέων για την Ευρώπη αυτή, όταν η Ευρώπη μόνο απόγνωση τους προσφέρει. Και γι' αυτό η σοσιαλδημοκρατική ομάδα απαιτεί ένα σύστημα εγγύηση τη κατάρτιση και τη απασχόληση για το νέο. Ο νέο θέλει Ευρώπη και δουλειά μέσα στην Ευρώπη. Μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα νέο που θα θέλει και την ίδια την Ευρώπη. Και επίσης ε, κοινωνική, κοινωνικό μοντέλο σημαίνει προστασία όλων εκείνων που βρίσκονται μέσα στην Ευρώπη και εκείνων που δεν έχουν γεννηθεί μέσα στην Ευρώπη και θεωρούνται ανάλογα με το σύστημα το δικαιικό ή το ένομο πει, Όλοι αυτοί πρέπει να χαίρουν των, ε, της προστασίας της κοινωνικής και μέσα στην Ευρώπη, για να μην κινδυνεύσει η κοινωνική μας ειρήνη. Πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν τους αποκλεισμού. Αντί για Βίλντερς, Λεπέν, νεοφασιστικά κόμματα στην Ελλάδα, Χρυσή Αυγή, πρέπει εμείς αυτούς τους νέους, αυτούς τους ξένους, αυτούς τους ε, μετανάστες να πούμε έχετε θέση εδώ στην Ευρώπη και μπορείτε μέσα στην Ευρώπη να αισθάνεστε στο σπίτι σας. Σε μια συζήτηση κυρίες και κύριοι που είχαμε χτες εδώ με νέους, ένας από τους ομιλούντες είπε αυτή η κρίση δεν είναι μια θεϊκή τιμωρία, δεν είναι σταλμένη από τον ουρανό, είναι μια τιμωρία την οποία εμείς οι ίδιοι φέραμε πάνω στα κεφάλια μας. Αυτή λοιπόν πρέπει να είναι και η απάντηση μαζί βέβαια, όλοι μαζί μπορούμε να πολεμήσουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και για να δώσουμε απαντήσεις σε αυτές τις δυνάμεις της καταστροφής, τις ακραίες δυνάμεις στην Ευρώπη. Όλοι μαζί, σοσιαλδημοκράτες ενωμένοι και Όλοι όσοι μίλησαν θετικά για την Ευρώπη πιστεύω πρέπει να δώσουμε τα χέρια για να στηρίξουμε αυτή την Ευρώπη που είναι για όλους μας και από όλους μας. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Σφόποντα. Τώρα εκ μέρου τη συμμαχία των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών ο κύριο Φερχόφστατ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα κι εγώ όσο ο κύριο Σφόποντα να παραφράσω αυτά που είπε ο νεοστή εκλεγής πρόεδρος στη Γαλλία, που είπε «Η αλλαγή είναι τώρα». Εγώ θα έλεγα απλώ η Ευρώπη είναι η αλλαγή και χρειαζόμαστε την Ευρώπη τώρα, στις 9 Μαΐου. Λαμβάνοντας υπόψη το πόσο σοβαρή είναι η κρίση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε γιατί Ωραία είναι να λέμε τόσα καλά πράγματα και τόσα καλά λόγια για το παρελθόν. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή κρίση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Η Ευρώπη περιθωρικοποιείται στον κόσμο. Η Ευρώπη αντιμετωπίζεται, αντιμετωπίζει μια συγκυριακή επιβράδυνση της οικονομικής τους ανάπτυξης και χρειάζεται να αντιμετωπίσει το γεγονό ότι την προφθαίνουν όλο και περισσότερο οι αναδυόμενε χώρε. Επίση, αντιμετωπίζει μια δημογραφική γύρανση. Η Ευρώπη είναι ένα κόσμο ο οποίο είναι πια πολύ πιο νέο και ο οποίο θα φτάσει σύντομα στα 10 δισεκατομμύρια κατοίκου. Η Ευρώπη είναι κατακαιρματισμένη, είναι διχασμένη μεταξύ των κρατών μελών της σε έναν κόσμο ο οποίος όλο και πέρα, όλο και πιο πολύ ενοποιείται αλλά και κυριαρχείται από τις μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, αντίθετα από αυτά τα οποία ισχυριζόμαστε, η κρίση αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Ευρώπη δεν είναι μια κρίση της παγκόσμιας οικονομίας. Ούτε καν μια κρίση των παγκοσμίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι μια ευρωπαϊκή κρίση και ιδίως μια κρίση των ευρωπαϊκών κρατών. Εδώ και κάποια χρόνια, πρέπει να το αναγνωρίσουμε σήμερα στις 9 Μαΐου, εδώ και πολλά χρόνια η Ευρώπη πλέει χωρίς πηξίδα, χωρίς ορίζοντα, χωρίς ελπίδα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορεί να βρει τη σωστή κατεύθυνση και να βρει λύσεις οι οποίες θα διαρκέσουν. Η 9, λοιπόν, 9η Μαΐου λοιπόν, αντί να είναι μια ευκαιρία για αυτοπανηγυρισμούς, για αμοιβαίους αμοιβαία συγχαρητήρια, θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε για την ανάγκη να δώσουμε μια νέα απάντηση σε αυτή την κρίση και όχι μονάχα με την πολιτική των μικρών βημάτων. Θα πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο ποιοτικό άλμα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε άρδιν αυτή την κατάσταση. Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύω ότι η Ευρώπη ή θα είναι ομοσπονδιακή ή δεν θα είναι, ή δεν θα υπάρξει πια. Αυτή είναι η επιλογή. Θα πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε τις λέξεις, να φοβόμαστε τη λέξη φεδεραλισμός για το μέλλον της Ευρώπης. Χρειάζεται μια φεδεραλιστική λύση στα προβλήματα της Ευρώπης που θα οδηγήσει σε μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση την οποία έχουμε ανάγκη. Ένα πραγματικό δημοκρατικό έλεγχο που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ένα πραγματικό ευρωπαϊκό θησαυροφυλάκιο, ένα ομοσπονδιακό προπολογισμό τη Ευρώπη και γιατί όχι, εν καιρό θα μας φέρει αυτό σε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό στρατό. Δεν έχουμε επιλογή. Το τονίζω, ο ευρωπαϊκός φεδεραλισμός είναι η μόνη λύση για να μπορέσουμε να ενσωματωθούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διαπραγματευόμαστε σαν ίσος προς ίσο. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διατηρήσουμε τον οικονομικό και πολιτικό ρόλο μας. Είναι ο μόνος τρόπος να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό υπόδειγμα. Πιστεύω επίσης κύριε Πρόεδρε ότι σήμερα στις 9 Μαΐου είναι και η στιγμή να γυρίσουμε σελίδα. Να ξεπεράσουμε τις ψευδεστήσεις μας. Τις ψευδεστήσεις εκείνων που θεωρούν ότι μόνο η λιτότητα θα μας βγάλει από την οικονομική κρίση αλλά και τις ψευδεστήσεις των άλλων που θεωρούν ότι η ανάπτυξη μπορεί να επανέλθει χωρίς να θέσουμε τάξη στα δημόσια οικονομικά μας. Είναι ένα μεγάλο λάθος λοιπόν αυτό το οποίο έχει γίνει τις τελευταίες χώρε να τεθούν αυτές οι δύο προσεγγίσεις ως αντιμέτωπε. Δεν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ της δημοσιονομικής πειθαρχία και της ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε και τα δύο. Και ανάπτυξη και λιτότητα και πειθαρχία αλλά και αλληλεγγύη. Αγαπητοί συνάδελφοι, το δημοσιονομικό σύμφωνο δεν πρέπει να αλλάξει θα πρέπει να προσθεθούν και άλλα στοιχεία στο Δημοσιονομικό Σύμφωνο και το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα πρέπει να αυξηθεί. Όλα τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία είναι στη διάθεσή μας θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Και τέλος, αυτά τα περιβόητα project bonds, αυτά τα ομόλεγα, πόσες φορές τα έχουμε συζητήσει εδώ στην αίθουσα. Και τέλο ε, πρέπει να έχουμε αυτό το κοινό ταμείο διάσωσης. Θα πρέπει να δώσουμε ε, τη δυνατότητα να πληρώσουμε τους ομολογιούχους ώστε να έρθουν νέα χρήματα και νέες επενδύσεις στην Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το μήνυμα για την 9η Μαΐου είναι πολύ συγκεκριμένο. Εάν εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να επιβιώσουμε, χρειαζόμαστε φεντεραλισμό. Ευρωπαϊκό φεντεραλισμό. Ο φεντεραλισμός δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φοβόμαστε. Είναι το μέλλον τη Υπήρου μα και το μέλλον ξεκινά σήμερα, την 9η Μαΐου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φερχόφστατ. Εκ μέρους των Πρασίνων Πράσινης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας, ο κύριος Κονπέντιτ. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, γκί, σε ευχαριστώ. Ίσως μπορέσουμε να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή, γιατί πιστεύω πράγματι ότι εάν μιλούμε για την 9η Μαΐου, αν μιλούμε για την Ευρώπη, αν μιλούμε για όλα τα επιτεύγματα, πρέπει να μιλούμε όμως και για αυτά τα οποία πρέπει ακόμα να επιτύχουμε για να έχουν ένα μέλλον οι Ευρωπαίοι πολίτες, για να τους ανήκει το μέλλον. Και δεν πρέπει ελαφρά την καρδία να κοιτάμε τα όσα συμβαίνουν σήμερα με τις εκλογές. Διότι εάν υπάρχει οικονομικό Εάν υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρώπη, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ε, εάν θέλουμε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, αυτή πρέπει να είναι δημοκρατική και αυτή πρέπει να είναι σε θέση να δίνει απαντήσει στα προβλήματα και του φόβου και τα άγχη των πολιτών. Κοιτώντα λοιπόν προ την Ελλάδα και τι εκλογέ που έγιναν εκεί σήμερα και όπου η μόνη λύση που βρήκε η Κεντρική Τράπεζα ήταν να πει δεν υπάρχει εναλλακτική στα όσα αποφασίστηκαν, τότε εγώ θα πω στην Κεντρική Τράπεζα προσοχή, προσοχή, Θυμηθείτε τι μας διδάσκει η ευρωπαϊκή ιστορία. Θυμηθείτε τι διδάσκει η ιστορία της Γερμανίας. Θυμηθείτε το σύμφωνο των Βερσαλιών. Όταν λέμε στους λαούς λύσεις δεν υπάρχουν, εναλλακτικέ δεν υπάρχουν, οι λαοί βρίσκουν εναλλακτικέ, οι οποίες είναι μερικές φορές αποτρόπες και γι' αυτό εμείς έχουμε ευθύνη και πρέπει να θυμούμαστε τι μας διδάσκει η ιστορία. Όταν στη δημοκρατία λέει κανείς δεν υπάρχει εναλλακτική, απαραίτητα ασφάλει. Η δημοκρατία πάντα συνεπάγεται αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Ιδάλως, καλύτερα να μην, να μην ασχολείται κανείς με την πολιτική. Και θα πω ένα πολύ απλό πράγμα. Εάν θέλουμε εάν δεν θέλουμε μάλλον η Ελλάδα να παρασυρθεί σαν ένα κικαιώνα επαναληπτικών εκλογών, μία, δύο, τρει, τέσσερι φορέ, μέχρι ότου φτάσει να πει συγγνώμη, συγγνώμη Ευρώπη, εξηλαιωθήκαμε και σα κάνουμε ό,τι θέλετε, τότε πρέπει να ξανανοίξουμε αυτό το μνημόνιο, πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το μνημόνιο, πρέπει να προτείνουμε κάτι στο λαό τη Ελλάδα. Γιατί αν δεν προτείνουμε τίποτα στους Έλληνες, οι προσεχείς εκλογικές αναμετρήσεις, θα δώσουν τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Το να αναθεωρήσουμε το μνημόνιο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Σημαίνει μόνο ότι πρέπει όντως ο λαός της Ελλάδας να μπορέσει να παρακολουθήσει, να είναι ικανός να παρακολουθήσει το ρυθμό των μεταρρυθμίσεων, να μην του στερήσουμε την ανάσα, την πνοή, το φαΐ, την τροφή και την, ε, το νερό. Γιατί αν τον φτάσουμε σε αυτή την ακραία κατάσταση θα δώσει ακραίως αντιδραστική, ναζιστική, σταλινιστική, ακραίως ακραία ακροδεξιά λύση. Στη Γαλλία ψήφισε ο γαλλικός λαός. Ξέρετε ότι είχα τοποθετηθεί και είχα μάλλον τοποθετηθεί υπέρ του ε, υποψηφίου που κέρδισε τις εκλογές. Αυτό όμως που δεν αντιλαμβάνομαι και δεν καταλαβαίνω σε αυτό που πράττουν οι άλλοι Ευρωπαίοι είναι ότι δεν είναι δυνατόν να λέτε στο γαλλικό λαό μετά από μια τόσο τεταμένη εκλογική αναμέτρηση δεν μπορείτε να του λέτε είτε είναι ο Λόντ είτε είναι ο Σαρκοζή αυτός που επιλέξατε, πάλι τα ίδια θα πρέπει να κάνετε. Γιατί τότε γιατί να κάνει εκλογέ ο λαό. Γιατί να πάει στην κάλπη ο λαό. Εάν σήμερα λοιπόν ο γαλλικό λαό σε μια πλειοψηφία που δεν είναι συντριπτική έστω και η κατάσταση θα είναι και δύσκολη αλλά ε, αποφασίζει παρόλα αυτά ότι θέλει να αλλάξει οφείλει ολόκληρη η Ευρώπη να αναλογιστεί πώς μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή. Και ο κύριος Μόντι, εάν έτεινε βικονούς στα μηνύματα που του στέλνει ο Ιταλικός λαός, γιατί τα είδαμε και τις δημοτικές εκλογές, θα πρότεινε κάποιες αλλαγές και στην Ιταλία. Και ο κύριος Ράχο στην Ισπανία πρέπει να προτείνει κάποιες αλλαγές, να καταλάβει ότι χρειάζεται αλλαγή και εκεί. Είναι προφανές λοιπόν ότι τώρα δεν είναι θέμα να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, σταθερότητα, ανάπτυξη κ.ο.κ πρέπει πλέον να δώσουμε ελπίδα στους λαούς της Ευρώπης. Αυτή την ελπίδα δεν μπορούν να τη δώσουν οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Εμείς οι Ευρωπαίοι, εμείς πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας και να γίνουμε φορείς της ελπίδας για, τον Ευρωπαϊκού για τους ευρωπαϊκούς λαούς, για τον Ευρωπαίο. Τι σημαίνει αυτό, ευρωπαϊκός προπολογισμό. ήδη η και σωστά λέει ο Γκί ότι πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, επενδύσουμε, ότι πρέπει να τη μετατρέψουμε σε ένα χρήσιμο εργαλείο, πρέπει να θεσπίσουμε ένα πρόγραμμα για ένα νέο πράσινο deal, για μια νέα πράσινη συμφωνία, μετατροπή δηλαδή οικολογική τη ευρωπαϊκή οικονομία που θα δημιουργήσει και θέσει εργασία. Και αν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό μέσω δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με ανάκαμψη τη οικονομία και μετά με τον προπολογισμό τον ευρωπαϊκό που θα έχουμε στη θέσή μα να, να επιστρέφουμε σιγά σιγά αυτό το δάνειο Εάν δεν το κάνουμε αυτό, εάν σταματήσουμε, εάν δεν εξασφαλίσουμε την ανάκαμψη ευρωπαϊκή οικονομία, εάν επαναπαυθούμε και πούμε θα δείτε, θα δείτε όλα θα πάνε καλά, οι νεοφιλελεύθερε οικονομίε όπω είδατε μα έφεραν με την πλάτη στον τοίχο και πρέπει να το πούμε, πρέπει να το φωνάξουμε σε όλε τι κυβερνήσει, εάν δεν αλλάξουν αυτού του ρυθμού του οικονομικού, όλοι θα βρεθούμε με την πλάτη στον τοίχο, αν όχι με το πρόσωπο. Και θα πω ένα πολύ απλό πράγμα. Ότι και οροφυλακτεί ένα τεράστιο κίνδυνο, ο οικονομικό, αλλά και ένα άλλο. Ο κίνδυνο για την ίδια τη δημοκρατία. Εάν πάψει να μα πιστεύει ο πολίτη, αν θεωρεί ότι πια δεν είμαστε ικανοί να χειριστούμε, να λάβουμε αποφάσει, να λάβουμε τι αποφάσει που χρειάζονται για τι αλλαγέ, τι απαραίτητε, τότε θα πάψει να πιστεύει ο λαό και αντί για μια επανάσταση που θα μας έδινε σε όλους μια λύση σωτηρίας θα μας οδηγήσει στη φρίκη η δημοκρατία που μας επιτρέπει να αποδείξουμε σήμερα ότι υπάρχει δυνατότητα επανεξισορροπήσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές, να θέσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό στο επίκεντρο, την Ευρώπη δηλαδή, στο επίκεντρο επακριβώς αυτής της απαραίτητης μετάλλαξης, ώστε να διαπιστώσει και ο πολίτης ότι ναι, είχε δίκιο όταν πριν από 60 χρόνια έχτιζε την Ευρώπη και πρέπει να του δώσουμε δίκιο για να κερδίσουμε και το μέλλον. Ιδάλλως το μέλλον θα το σφετεριστούν οι αγορές και θα διώξουν από αυτό τον, τους λαούς της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κονβεντίτ για την συντηρητική και μεταρρυθμιστική ομάδα. Ο κύριος Κάλανεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Σουμάν, ο Μονέ και ο Σπινέλη έζησαν σε μια τελείως διαφορετική Ευρώπη από τη σημερινή και η Ευρώπη, η Ήπειρός μας, ε, ε, έζησε δύο παγκόσμιους πολέμους και η πρόκληση τότε ήταν να υπάρχουν τρόφιμα στο τραπέζι. Και υπήρχε ένας τείχος το οποίο ε, διαιρούσε το Βερολίνο παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, η κοινή γεωργική πολιτική και τότε οι πολιτικές αυτές μας επέτρεψαν να επιτύχουμε κάποιους από τους στόχους. Διεύρυνση προς Ανατολής, ε, η οποία έφερε ελευθερία ε, στους ανθρώπους και πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. Αλλά κυρίες και κύριοι, άλλαξε ο κόσμος ε, πολύ από τότε που έγινε η δήλωση του Ρομπέρ Σουμάν. Σε πολλού τρόπου όμω η Ευρώπη δεν έχει αλλάξει. Πολλέ από αυτέ τι καινοτόμε λύσει τη εποχή έχουν γίνει τμήμα του προβλήματο του 21ου αιώνα. Και η Ευρώπη γίνεται αδιάφορο όχι μόνο για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και στο μυαλό πολλών πολιτών μα. Και να σα πω ότι Οι πολίτε δεν εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμπιστεύεται του πολίτε. Η δημοκρατία, ο κανόνα των ανθρώπων είναι η το μεγαλύτερο εξαγώγημο προϊόν τη Ελλάδο και είναι αυτή τη στιγμή που απειλεί. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, οι όροι της Τρόικας, ε, η ΑΕΝΑ, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν επιτρέπουν στους πολίτες μας να μπορούν να καθορίσουν τη μοίρα τους και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να θεωρούμε τους ανθρώπους δεδομένους. Εάν συνεχίσουμε να φερόμαστε έτσι θα στραφούν σε αποτρόπες αναλλακτικέ λύσεις, σε κομμουνιστές και νοναζί που θέλουν ε, να θέσουν φράχτες στα ελληνικά σύμμορα και δυστυχώς ε, τώρα αποτελούν και τμήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ε, η κυρία Λεπέν έλαβε το 1 πέμπτο των ψήφων στη Γαλλία. Και τι βλέπουμε από τα αποτελέσματα στη Γαλλία. Κάποιος μας είπε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό συνοψίζει όλα όσα είναι στραβά με την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στη δήλωση αυτή. Η δήλωση του Σουμάν υποστηρίζει ακριβώς αυτή την υπόθεση. Είχαμε πολύ καλές προθέσεις, οι οποίες όμως έγιναν τμήμα του προβλήματος και δεν αφήνουν πλέον καμία δυνατότητα οικονομικής ελευθερίας στους ανθρώπους να παραφιάσω μια διάσημη φράση του Πρόεδρου Ρίγκαν. Εγώ είμαι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Εγώ πιστεύω ότι μια μικρή κυβέρνηση βοηθάει. Όταν οι εθνικές κυβερνήσεις ε, ε, είδαν τι γίνεται με τα κράτη, κατάφεραν να έχουν ε, αποτελέσματα στην οικονομία και η Ευρώπη δυστυχώς έγινε μια μεγάλη κυβέρνηση και πρέπει να υπαναχωρήσει τώρα στα σύνορά της. Κάποιοι είπαν ότι οι εκλογές της Κυριακής ήταν ε, η νίκη των πολιτικών που αντικατέστησαν αυτούς που είναι υπέρ της λιτότητας. Αυτό βέβαια είναι λανθασμένο. Οι περισσότεροι από όσους γνωρίζω, ίσως με την εξαίρεση των πρασίνων, επιθυμούν την ανάπτυξη. Η βιώσιμη ανάπτυξη όμως απαιτεί κατάλληλη παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σήμερα. Και θα πρέπει να δαπανούνται περισσότερα ε, χρήματα για να δημιουργηθούν ψευδείς ε, ε, ζητήσεις και αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ανάπτυξη είναι βλακώδες, δεν είναι βιώσιμο και θα φτάσουμε πολύ πιο κοντά στην εθνική χρεοκοπία για περισσότερα κράτη-μέλη. Η πολιτική μου ομάδα προσφέρει ένα λακτικό όραμα, το οποίο βασίζεται στην ελευθερία, στην εθνική δημοκρατία και στην κατάλληλη ανάπτυξη μέσω επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι το εμπόριο είναι ο καλύτερο τρόπο να προάγουμε την ανάπτυξή μα. Πιστεύουμε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι μικρότερος, θα πρέπει να δοθούν νέες προτεραιότητες στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, όπως για παράδειγμα η έρευνα. Πιστεύουμε στην ενιαία αγορά. Πιστεύουμε ότι η ενιαία αγορά είναι το μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να προάγουμε την έλλειψη νομοθεσίας και όχι τη γραβειοκρατία και την υποχρεωτική εναρμόνιση. Πριν από 7 χρόνια, μετά από την απόρριψη από πλευρά Ολλανδίας και Γαλλίας του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, ένας από τους ε, πολίτες του Στίβεν Χιούς ε, και από τη δική μου την επικράτεια, ο Τόνι Μπλερ, είπε ότι οι πολίτες ε, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου στα τείχη της πόλης, εμεί τίνουμε δίκονου. Ξέρουμε όλη την απάντηση. Αλλά πλέον ακούγεται πολύ πιο δυνατά ο θόρυβο από ό,τι ακούστηκε το 2005. Και θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσον εμεί τίνουμε δίκονου στο αυτό που έχουν να πούν οι πολίτες στη σημερινή ημέρα. Διότι οι πολίτε αντιμετωπίζουν ξεκάθαρες προκλήσει. Μπορούμε να περάσουμε περισσότερη νομοθεσία, μπορούμε να έχουμε δεκαετή προγράμματα, μπορούμε να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία όμω και να άρουμε το άχθο για τι επιχειρήσει. Να εξακολουθήσουμε να φρονούμε ότι εμεί είμαστε που γνωρίζουμε τι είναι το σωστό, ενώ θα μπορούσαμε και να επιτρέψουμε στου πολίτε να γνωρίζουν αυτοί ποιο είναι το σωστό. Θα πρέπει να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει λιγότερα αλλά τα κάνει καλύτερα. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, να αναγκαλίσουμε τι μικρέ κυβερνήσει στην Ευρώπη. Ο χρόνο περνάει και αν δεν αλλάξει ο κόσμο, ε, ο κόσμος ούτως ή άλλως θα συνεχίσει να γυρίζει και η Ευρώπη θα μείνει ε, στην ε, ε, τελευταία σειρά ουραγός όλου του υπόλοιπου κόσμου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κάλνεν. Ο κύριος Φάρατς για δύο μισή λεπτά. Well, happy Day. Χρόνια πολλά. Χαρούμενη ημέρα της Ευρώπης, η ημέρα Σουμάν. Νομίζω ότι έχουν σιωπήσει όλοι οι πανεγυρισμοί. Μόνο ο κύριος ε, Σούλτς εδώ ε, μας ε, χρησιμοποίησε τα αγγλικά και θριαμβολόγησε. Όλοι αναφέρονται στην επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι δεν λέει κανένας ότι δεν το πιστεύει κανείς πλέον αυτό δεν θα έπρεπε να γιορτάζουμε την 9η Μαΐου, θα έπρεπε να γιορτάζουμε την 8η Μαΐου, την ημέρα της συνθηκολόγησης στην Ευρώπη και της νίκης. Την τελευταία ημέρα που οι Γερμανοί προσπάθησαν να κατακαιρματίσουν την Ήπειρο και τα κατάφεραν και οι περισσότερες χώρες της Ήπειρου έλαβαν πάλι πίσω τη δημοκρατία τους. Ενώ στις 9 Μαΐου γιορτάζουμε μια άλλη προσπάθεια να πατάξουμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Ε, δεν πιστεύω ότι είχε καλές προθάσεις ο Ζαμονέ. Πίστευε ότι αν καταργήσει τα κράτη-έθνη δεν θα μπορούσε να είχε άλλο πόλεμο. Αλλά βέβαια τότε δεν μπορούσε να δει πώς ε, ε, θα διαδραματιστεί η θεωρία του στη Γιουγκοσλαβία. Και βέβαια, όπως με όλους τους πολέμους, ε, πήγανε πολύ άσχημα τα πράγματα και πλέον ο Ευρωπαϊκός Τιτανικό έχει χτυπήσει το παγόβουνο. Έχουμε οικονομική χρεοκοπία, ε, έχουμε ανεργία, αλλά κυρίως έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με την οικονομική φυλακή του ευρώ, η οποία αποτελεί πλέον τεράστιο κίνδυνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να υπάρχει μαζική αναταραχή, μπορεί και επανάσταση σε κάποιες χώρες οι οποίες οδηγούνται στο χείλος της απελπισίας. Υπάρχει όμως ίσως μια ευκαιρία, ίσως κάποια καλά νέα. Μπορεί πλέον να έχει ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή επανάσταση, μια δημοκρατική επανάσταση. Ξεκίνησε στη Φιλανδία ε, πέρσι όπου είχαμε νέα πολιτικά κινήματα ε, της... Ε, ε, άκρα δεξιά ή τη αριστεράς να έχουν καλά αποτελέσματα. Αλλά δεν έχουμε πάντα καλά αποτελέσματα. Αυτό που είδαμε στην Ελλάδα την περασμένη Κυριακή θύμισε λίγο τη Γερμανία του 1932. Έχουμε πλέον τα άκρα να επικρατούν και αυτό μπορεί να οδηγήσει και στην αναγέννηση του εθνικοσοσιαλισμού στην Ευρώπη. Οδεύουμε προς τη λανθασμένη κατεύθυνση και θα πρέπει να σταματήσουμε την Ευρωζώνη, θα πρέπει να απελευθερώσουμε τις χώρες της Μεσογείου και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη. Και εγώ θέλω Ευρώπη, αλλά μια Ευρώπη θα βασίζεται στο εμπόριο, στη συνεργασία, στο γεγονός ότι θα καθίσουμε όλοι γύρω από ένα τραπέζι και θα συμφωνήσουμε για συγκεκριμένους κανόνες για να προστατεύσουμε το περιβάλλον για οτιδήποτε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, αλλά όχι πίσω από αυτή τη σημεία. Εγώ δεν πρεσβεύω σε αυτή τη σημεία και οι περισσότεροι πολίτες ούτε και αυτοί πρεσβεύουν σε αυτή τη σημαία. Ευχαριστώ κύριε Φάρατς. Ο κύριος Λεγιαρή και τρία λεπτά έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου για τον φόρο τιμής που απέτησε στο συνάδελφό μας Μιγγέλ Πόρτας πριν από λίγο. Ο Πρόεδρος έκανε μια πραγματική ε, ένα έπαινο της Ευρώπης, αλλά αυτά δεν αποτελούν πραγματικότητα. Αν υπάρχουν τόσο μεγάλοι κίνδυνοι κατάρρευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είναι χωρίς κατεύθυνση πολιτικοί ηγέτες, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Η λιτότητα έκανε το, τους λαούς να προχωρήσουν σε εξαναγκαστική πορεία. Όλο και περισσότερο ιδιωτικοποιούνται τα δημόσια αγαθά και οι πολιτικές παρόλα αυτά δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και πολύ γρήγορα. πρέπει να καταλάβουμε τι έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Το Ρουμανικό Κοινοβούλιο ανέτρεψε το σχέδιο ε, νίκη της, ε, του Ολάντ στην, ε, στην Γαλλία. Νίκη στις ε, τοπικές εκλογές της αντιμνημονιακής πτέρυγας. Στην Ελλάδα επίσης νίκη των αμνομονιακών. Θα πρέπει λοιπόν να ξεχάσουμε το memorandum της Τρόικα και να βρεθεί ένας νέος δρόμος στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες. Θα πρέπει να ξεχάσουμε τη λιτότητα του Σαρκοζή και της Μέρκελ και το λεγόμενο πρωτόκολλο ανάπτυξης που είναι αντίθετο στις ίδιες τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να το εγκαταλείψουμε και να βρούμε ένα άλλο δρόμο. Θα πρέπει να βρούμε ένα νέο σύμφωνο ανθρώπινης, οικολογικής και κοινωνικής ανάπτυξης με νέο ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία πρέπει να δώσει πιστώσεις για την ανάπτυξη, για τη βελτίωση της αγοραστικής δύναμης, για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της απασχόλησης, για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, τις δημόσιε υπηρεσίες και την οικολογική μεταλλαγή της υπήρου μας ένα τελείω διαφορετικό λοιπόν μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τη οποία το κεφάλαιο θα πρέπει να αυξηθεί, η καλύτερη χρήση των διαρθρωτικών πόρων, ο φόρο για τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ, ένα φόρο εναρμονισμένο για τα κεφάλαια, θα είναι λοιπόν ο μοχλό που θα οδηγήσει σε αυτή την ανθρώπινη ανάπτυξη, στην οποία πρέπει να προσθέσουμε την δημιουργία χρήματο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προ όφελο των κρατών και όχι μονάχα των τραπεζών. Θα πρέπει να αποφύγουμε <clears throat> τον λανθασμένο ανταγωνισμό με ένα ελάχιστο εισόδημα και ελάχιστες αμοιβέ στην Ευρώπη μαζί με ένα ε, σχέδιο δράσης κατά της ένδυας. Θα πρέπει να έχουμε ένα μορατόριο για τα χρέη του παρελθόντο και θα πρέπει να ζητάμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να δανείζει τα κράτη με 1% επιτόκιο όπω στις Τράπεζε. Θα ήθελα η Κομισιόν και το Συμβούλιο να μας δώσουν εκθέσεις για τη χρήση του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει δανείσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ιδιωτικές τράπεζες. Και επίσης ενώπιον των προκλήσεων και των απειλών που έχουμε ενώπιον μας, θα πρέπει το Κοινοβούλιο να πάρει την πρωτοβουλία ενός μεγάλου Ευρωπαϊκού Φόρουμ με συμμετοχή όλων των, Ευρωπαϊκών, των Εθνικών Κοινοβουλίων με τις ενώσεις των πολιτών, τα συνδικάτα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια πλήρη αναδιάρθρωση και μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λεγιαρίκ. Ακροκολουθεί και ο Σώσα Βάγνερ για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είδαμε να εκτιλήσετε μια μεγάλη διαμάχη που έχει να κάνει με τις αντίμαχες έννοιες της λιτότητος και της ανάπτυξης. Από αυτά που ακούσαμε φαίνεται ότι η ιδέα της ανάπτυξης είναι μια επινόηση των τελευταίων ημερών. Αυτό είναι πολύ μακριά <clears throat> από την πραγματικότητα. Έχει ξεκινήσει το 1997 από το σχέδιο ανάπτυξης και σταθερότητας. Και η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική έρευνα είναι πολιτικέ οι οποίε συνεχίζουν την ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών. Και ε, απευθύνομαι προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη του Κοινοβουλίου που έχουν τη δυνατότητα να εισακουστούν ε, εμείς δεν έχουμε κανένα σύμπλεγμα όταν θα γίνει η συγκεκριμένη συζήτηση. Εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με ψηλά το κεφάλι και αυτή είναι η άποψή μου, μειονοτική μεν, αλλά μεταξύ των εγγεγραμμένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δεν επιτρέπεται το χειροκρότημα από τα θεωρία των επισκεπτών. Δεν ανήκει στις παραδόσεις τη κοινοβουλευτική. Και τώρα